Genau. So. Good morning. Good morning. Good morning. Καλημέρα σας. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος. Εδώ, σήμερα, θα ήθελα ως πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίου Ελέγχου να καλωσορίσω τα μέλη της Επιτροπής των Προπολογισμών που ήρθαν για αυτήν την κοινή συνεδρίαση που θα αφορά τον κανονισμό επί του προϋπολογισμού. Και πρώτα πρώτα θα δώσω τον λόγο στον, στην κυρία Χάουγ για την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ. Την κυρία Χάουγ. Η σημερινή συνεδρίαση είναι αποτέλεσμα εντατικών εργασιών και διαπραγματεύσεων που είχαμε με το Συμβούλιο. Τελικά απέδωσαν καρπούς αυτές οι επαφές και μόλις σήμερα το πρωί είχαμε και κάποια από τα αποτελέσματα. Επιθυμούμε δεν να διεξαγάγουμε μία μόνη ψηφοφορία. Δεν έχουμε ήδη να κάνουμε τόση πολλή ε, δουλειά πια, διότι έχει ήδη ολοκληρωθεί και ευχαριστώ εδώ τους κυρίους, ε, την κυρία Γκρέσλε και τον κύριο Ριβελίνη και συγχαίρω επίσης τα πρόσωπα αυτά για τις ημέρες, εβδομάδες, μήνες ε, εργασίας που έχουν καταβάλει. Διότι είχαμε ακούσει, έχουμε ακούσει μάλλον και τις εκθέσεις τους σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και προσπαθήσαμε, προσπαθήσαμε επαναλαμβάνω, να κινηθούμε με την ίδια ταχύτητα όπως η διαπραγματευτική ομάδα. Ελπίζω ότι το καταφέραμε και φτάνουμε πια στο αποκορύφωμα με των προσπαθειών μας. Λέω αποκορύφωμα εννοώντας ότι αρχίζουμε και βλέπουμε την κορυφή. Ευχαριστώ λοιπόν αγαπητοί Ινγκεμπόργκ, ευχαριστώ κύριε Ριβελίνη και σας χειροκροτώ. Äh, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Χάουκ. Ως ας πούμε ελεγκτής του προϋπολογισμού είμαι άνθρωπος νυφάλιος και θα εκφράσω τη χαρά μου όταν θα δω να έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα, λέει ο κύριος Τόερερ. Ευχαριστώ και ε, συμφωνώ με τα συγχαρητήρια προς τους δύο εισηγητές διότι είναι αναρρύθμιτες οι διαβουλεύσεις, οι τριμερείς διάλογοι και ούτω καθεξής. Πριν όμως αρχίσουμε να ζητοκραυγάζουμε, απευθύνω χαιρετισμό και στους εκπροσώπους του Συμβουλίου που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσά μας, θα πρέπει να δούμε πού πρέπει να κινηθεί το Κοινοβούλιο για να καταλήξει σε μια κοινή βάση, διότι έχουμε αποσυνδέσει έναν αριθμό πραγμάτων που ωστόσο συνδέονται με το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η συμβαστική λύση λοιπόν που επιτεύχθηκε αποτελεί όντως πρόοδο, είναι αξιοπρεπής και εννοώ επί της ουσίας, δηλαδή για την καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Μακάρι να είχαμε επιτύχει περισσότερα θα τα ακούσουμε, θα τα αξιολογήσουμε, θα τα συζητήσουμε, θα ψηφίσουμε μετά. Πρόκειται για ψηφοφορία που ε, βρισκόμαστε απέναντι στο δίλημα ή τρίλημα υπέρ, κατά και αποχές. Υπάρχουν και γνωμοδοτήσεις τις οποίες έχετε λάβει, έχουν διαβιβαστεί σε όλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτός και αν όχι θα σας τις πω ώστε ο καθένας να έχει τη δυνατότητα να τις λάβει υπόψη του. Προβλέπετε λοιπόν 23 Οκτωβρίου Τρίτη στην περίοδο συνόδου η ψηφοφορία εφόσον δεν αλλάξει τίποτε επ' αυτού εφόσον ψηφιστεί θα έχει προχωρήσει ένα σοβαρό νομοθέτημα, θα έχει ολοκληρωθεί λοιπόν, που οφείλουμε όπως είπα στην προεργασία των κυρίων Ριβελίνη και Γκρέσλε, που την σημασία της δουλειάς τους την τονίζω και πάλι, διότι η συνεργασία με την Ινκεμπορ Γκρέσλε στις διαπραγματεύσεις αυτές που ήταν αρκετά δύσκολες ήταν εξαιρετική. Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ανέλαβε η ίδια είναι και πολλή δουλειά, χωρίς την οποία δεν θα τα είχαμε πετύχει τα πράγματα αυτά έτσι. Τους ευχαριστώ, τους δύο και ρωτώ αν επιθυμούν να λάβουν το λόγο. Πρώτα ο κύριος Ριβελίνη. Αν θέλει. Α, η κυρία Κρέσλε θέλει να αρχίσει. Έχετε το λόγο κυρία Κρέσλε Όταν όλοι μου λένε καλά λόγια αρχίζω και δυσπιστώ. Φτάνουν τα καλά λόγια. Ευχαριστώ πολύ τον συνεισηγητή μου, καθώς και όλες και όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ βέβαια και τον πρόεδρο που διήφθηνε τους τριμερείς διαλόγους, καθώς και την κυρία Ιβάνοβα δίπλα μου. Ευχαριστώ και πολλούς επιμελείς ανθρώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που δούλεψαν όλο το καλοκαίρι για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Ευχαριστώ και για την ενθάρρυνση που μας δώσατε. Θέλω να γίνει και μια συζήτηση στην Ολομέλεια όπου να εξηγήσουμε τι πετύχαμε υπέρ των πολιτών, υπέρ της Ευρωπαϊκής Διοικήσεως και υπέρ των διοικήσεων των χωρών μελών. Πρόκειται και για μια απόδειξη ότι οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να συνεργαστούν εν τέλει χωρίς η μια να εμποδίζει το έργο της άλλης. Θα έρθω σε ένα σημείο, υπάρχουν αυτά τα draft statements, τα οποία έχουν προσαρτηθεί, υπάρχουν και κοινά statements και υπάρχουν και μονομερεί δηλώσεις δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τις μονομερείς δηλώσεις, ποτέ δεν τέθηκε θέμα να αποτελέσουν τμήμα του συνολικού κειμένου. Εγώ θυμάμαι τη συζήτηση, διότι εγώ είχα τότε δηλώσει ότι θα έβαζα να τα πει όλα αυτά το Συμβούλιο σε μονομερείς δηλώσεις. Αυτό ακριβώς για να δείξω πού μπορούν να καταλήξουν αυτές οι μονομερείς δηλώσεις. Μονομερείς δηλώσεις δεν έγιναν ποτέ δεκτές. Ούτε επιτρέπεται να προκαλέσουμε την εντύπωση δημοσιεύοντάς τις μαζί με το κοινό κείμενο να δώσουμε λοιπόν την εντύπωση ότι αποτελούν τμήμα του. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ σύμφωνοι με, την, με τις μονομερείς δηλώσεις. Τώρα υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θα συμπληρωθεί και γραπτός τα 85,9 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε το Βέλγιο στο Κοινοβούλιο για τα κτίρια. Το ποσό αυτό εξακολουθούμε να το, να το θεωρούμε external assigned revenue, εξωτερικό, εκ των έξωθεν προερχόμενο έσοδο. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αλλιώς τα χρήματα αυτά που πρέπει να εξοικονομήσουμε τα επόμενα χρόνια για τα κτίρια του Κοινοβουλίου, μετά από τις αλλαγές του δημοσιονομικού κανονισμού, επιστρέφουν στις χώρες μέλη. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε κάτι τέτοιο και γι' αυτό καταθέτουμε εδώ σε δήλωση την νομική μας άποψη. Το θέμα αυτό κάποια στιγμή ήταν δύσκολο να το διαπραγματευτούμε. Μαζί με την κυρία Χολμάιερ έχουμε κάνει ορισμένες πολύ καλές τροποποίησεις και δύσκολα μάλιστα Αυτό το ποσό λοιπόν, των 85,9 εκατομμυρίων από το Βέλγιο, θα υπαχθούν ακόμα, θα υπαχθεί υπό το παλαιό καθεστώς. Νομίζω λοιπόν ότι το αποτέλεσμα είναι καλό και είναι σημαντικό το καλό αυτό αποτέλεσμα να μπει και στον τομεακό κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρέσλε. Εσείς κύριε Ριβελίνη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να προσθέσω και πολλά άλλα σε αυτά που είπε η Σνέλφος Γκρέσλερ, πέραν του, των ευχαριστειών που θα ήθελα να απευθύνω προς όλους. Ε, επιτρέψτε μου όμως να κάνω μια πολιτική αξιολόγηση. Αυτή η μακρά εργασία είχε σαν κεντρικό στοιχείο την προστασία του Κοινοβουλίου από την κυρία Γκρέσλερ και ήταν πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι βρέθηκε μια συνέργεια μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων έτσι ώστε να δοθεί μια όθηση ε, στις ευρωπαϊκές πολιτικές σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ε, και δεν αναφέραμε μονάχα στις θέσεις του Κοινοβουλίου, αλλά και ε, προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες, πάρα πολλοί συμβιβασμοί. Και αυτή η εργασία που δεν είναι εργασία μόνο κοινοβουλευτική, μόνο ορισμένων ατόμων, αφορά όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί είναι πραγματικά αποτέλεσμα ενός, ε, μιας μεγάλης συνέργειας και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερο την Ίγκε. Είναι μια εξαιρετική γυναίκα, ένας σκληρός βράχος που νομίζω ότι <laughs> τη βλέπουν στα όνειρά τους εντός εισαγωγικών και το, και το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τις ε, απόψει των εισηγητών. Κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο. Αν θέλετε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία. Α, μισό λεπτό. Διαπρο... ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ πολύ. είναι σημαντική η ψηφοφορία και θέλω να ξέρω εάν οι κανόνες της πολυγλωσσίας έχουν γίνει ε, έχουν προστατευτεί. Γιατί διαφορετικά θα ήθελα κυρία Πρόεδρε και κυρία Πρόεδρε να υποβάλω ένσταση. Μπορούμε να διευκρινίσουμε το θέμα αυτό. Άμα δεν έχει τότε θα την ρίξει την Ε? Ο πρόεδρος κ. Στόλερ με ενημερώνουν μόλις ότι είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να ψηφίσουμε το ολοκληρωμένο κείμενο στα αγγλικά. Υπάρχουν βέβαια ορισμένες μεταφράσεις οι οποίες εξετάζονται από τους γλωσσομαθείς νομικούς και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ακόμα σε όλες τις γλώσσες αυτή η μετάφραση. Έχει λοιπόν δίκιο στην ένσταση του ο κύριος Οντί. Σημειώνουμε την ένσταση στο πρακτικό, αυτή είναι η πρότασή μου, και προχωρούμε στην ψηφοφορία, διότι αλλιώς δεν θα προλάβουμε λόγω του χρονοδιαγράμματος. Είναι όμως σημαντικό να τονιστεί η σημασία του γλωσσικού καθεστώτος. Βέβαια τα γεγονότα μας ε, πιέζουν και μας αναγκάζουν να προχωρήσουμε. Βέβαια, στην Ολομέλεια θα υπάρχουν όλες οι μεταφράσεις για την ψηφοφορία. Προτείνω λοιπόν, εάν συμφωνείτε με αυτή την σημείωση στο πρακτικό, να δηλώσουμε ότι έχουμε λάβει υπόψη την ένσταση αυτή, προχωρούμε στην σύσταση των δύο επιτροπών που είναι απαραίτητο να ψηφιστούν για να μπορέσει να ψηφίσει η Ολομέλεια είναι σημαντικό βεβαίω στην τελική ψηφοφορία να τηρηθεί απολύτω το γλωσσικό καθεστώ και εδώ με διαβεβαιώνουν ότι αυτό θα συμβεί. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, από την Επιτροπή Προπολογισμών είναι 11 τα μέλη. Διακόπτει ο πρόεδρος. Υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός. Υποθέτω ότι είναι παρόντα τα μέλη και οι αναπληρωτές τους η ψηφοφορία θα γίνει ηλεκτρονικά. Γι' αυτό θέτω το ερώτημα ποιος είναι υπέρ του συμβαστικού κειμένου για τον δημοσιονομικό κανονισμό, για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως υποβλήθηκε στα μέλη στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, καθώς επίσης και υπέρ των κοινών γνωμοδοτήσεων για το MFF, για τα κτίρια και για το άρθρο 195 παράγραφος 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Είναι ηλεκτρονική βεβαίω, είναι ονομαστική η ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρας τη ψηφοφορία. Διαπιστώνω ότι πρόκειται για σαφή πλειοψηφία και των δύο επιτροπών. Δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά βέβαια. Και πάλι συγχαρητήρια και από μέρος μου στους δύο εισηγητές για το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα και το καθαρό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ε, κυρία Χαουκ, ευχαριστούμε όλες και όλους τους συναδέλφους που προσήλθαν για να ψηφίσουν και καλή σας μέρα. Θα κάνουμε μια μικρή ε, ε, παύση πέντε λεπτών και θα συνεχίσουμε με τις εργασίες μας. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας. Der Bericht äh, von der Frau Hohlmeier haben wir vertagt, deshalb heute Αναβάλαμε την ε, μελέτη της έκθεσης της κυρίας ε, Μόνικα ε, Χολμάιερ και επομένως περνάμε αμέσως στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως που είναι το σημείο 13, δηλαδή μία μελέτη σχετικά με το πώς εποπτεύουν και ελέγχουν τους προϋπολογισμούς τους στα Εθνικά Κοινοβούλια. η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να έχει πιο στενές επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πολύ στον έλεγχο του προϋπολογισμού. Σας θυμίζω την ακρόαση που είχαμε πριν από λίγο καιρό για το USN ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τότε αγωνιστεί μαζί με κάποια εθνικά κοινοβούλια έτσι ώστε ε, να μπορεί να γίνει έλεγχος ε, των εθνικών λογαριασμών. Επομένω, ε, η αγαστή συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια είναι πολύ θετικό. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γκερμπράντι που είναι ο εισηγητή και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο πρώτα να έχουμε την παρουσίαση τη ίδια τη μελέτη και μετά. Προεδρο, απλώ ήθελα να σα δώσω την δυνατότητα να κάνετε κάποιε εισαγωγικέ παρατηρήσει εάν το επιθυμούσατε βεβαίω. Θα το κάνετε μετά. Πολύ ωραία. Επομένως θα δώσουμε το λόγο αμέσως ε, ε, στην κυρία Λόπες Φερνάντες, την καλωσορίζουμε μάλιστα που είναι εδώ μαζί μας και τον κύριο Μισό και θα τους δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Ε, λέει ο κύριος Χάμερ. Χθε το βράδυ είχαμε ωραίο καιρό, σήμερα έβρεξε όμως το πρωί, ελπίζω να μην είναι ε, ενδεικτικό του κλίματος που θα επικρατήσει όταν θα μιλάμε για το θέμα. Ε, είμαι εδώ μαζί με την κυρία Λόπες και δουλεύουμε μαζί για αυτήν την έκθεση, αυτήν την μελέτη. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω κάποιες ε, κάποιες πρώτες ε, παρατηρήσεις ε, για να σας πω ε, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία, στα οποία έχουμε καταλήξει. Τα κύρια στοιχεία ε, της ε, μελέτης αφορούσαν την αποτελεσματικότητα με την οποία δίνουν απαλλαγή ε, στους προϋπολογισμούς τους τα κοινοβούλια και θεωρήσαμε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλό να το γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν αναπτύσσει την δικιά του διαδικασία απαλλαγής και επίσης θεωρήσαμε ότι καλό ήταν να κάνουμε και κάποιες συστάσεις γύρω από αυτό το θέμα. Ε, επίσης το θέμα της αποτελεσματικότητας είναι σημαντικό. Πώς ορίζεται η αποτελεσματικότητα. Ξεκινήσαμε συζητήσεις με μέλη της διοίκησης του Κοινοβουλίου ε, ξεκινώντας από την διαπίστωση ότι από τη μία πλευρά πρέπει να μιλάμε για υγιή ε, και σωστή οικονομική διαχείριση, δηλαδή που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα ε, που θεωρούνται διεθνώς ως αποδεκτά ε, και από την άλλη πλευρά ότι καλύπτει τον ρόλο που παίζει σαν θεσμικό όργανο. Η προσέγγιση που επιλέξαμε ήταν να έχουμε μία ε, σύντομη έποψη όλων των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της διαδικασίας απαλλαγής και μετά ε, κάναμε 10 ε, μελέτες περιπτώσεων και ιστάτης από, ειδικές, από άλλες χώρες συν μία στην οποία περιλάβαμε ορισμένες ε, χώρες, ε, δηλαδή ε, Τσεχία, Γερμανία, Δανία, Εστονία, Φιλανδία, Γαλλία, συν Καναδά σαν μια εξωτερική χώρα. Ήταν σημαντικό για μας να κάνουμε και μία επιπλέον μελέτη περιπτώσεως και επιλέξαμε το καναδέζικο σύστημα. Επίσης κάναμε και μία έρευνα όσον αφορά το feedback των εμπλεκομένων μερών ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί μιλήσαμε με κοινοβουλευτικούς, κοινοβούλια κτλ. Και βεβαίως καταλήξαμε ε, στην συγκριτική ανάλυση. Αυτό που κατέστη προφανές άμεσα ήταν ότι υπάρχουν διάφορες προκλήσεις ε, στην διαδικασία της της ε, απαλλαγής. Δηλαδή ότι οι κοινοβουλευτικές δαπάνες δεν κατηγοριοποιούνται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ε, βλέπετε ας πούμε στην τρίτη στήλη, την περίπτωση της Γερμανίας δηλαδή, στο κάτω μέρος με το βαθύ γαλανό είναι ε, ε, ε, αυτό το οποίο πληρώνει η διοίκηση προς τρίτους ενώ ας πούμε στη Δανία το ποσοστό είναι τελείως διαφορετικό δηλαδή και το διοικητικό κόστος είναι διαφορετικό και δεν είναι εύκολο να πει κανείς ποιο σύστημα είναι το καλύτερο γιατί οι διάφορες διοικήσεις και οι κοινοβουλευτικές άρα διοικήσεις, διοικήσεις των διαφόρων κοινοβουλίων λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και επομένως δεν είναι εύκολο με τέτοιες διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις να προχωρήσει κανείς σε μια αποτελεσματική ε, συγκριτική ανάλυση γιατί τα στοιχεία διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επίσης μην λησμονούμε ότι ε, η κάθε χώρα έχει διαφορετικές παραδόσεις και ε, οι ιστορικές ε, διαδικασίες από τις οποίες γεννήθηκαν τα κοινοβούλια και οι τρόποι λειτουργίας τους διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Νομίζω ότι εδώ θα στραφώ προς την Κάρμεν και θα επανέλθω εγώ αργότερα με κάποιες συστάσεις και κάποια τελικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα που μας απασχόλησαν ε, ήταν ε, η ανάγκη ε, ταυτοποίησεων στη διαδικασία της απαλλαγής. Βλέπετε λοιπόν και την, την ανάγκη μεταρρύθμισης. Είναι ευπρόσδεκτη η ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, και εδώ σας δείχνουμε ένα γράφημα το οποίο δείχνει την, ε, το ποσοστό ε, της αποτελεσματικότητας έτσι όπως την καταλαβαίνουν τα ίδια τα κοινοβούλια και έτσι όπως την αναφέραμε και εμείς προηγουμένως, δηλαδή καλή διαχείριση και διαφάνεια. Με τον τρόπο αυτό η ακεραιότητα της διαδικασίας απαλλαγής μπορεί να συμβάλλει ε, στην δημιουργία καλής ε, λογοδοσίας ε, και ορθής αξιοπιστίας του Κοινοβουλευτικού Ιδρύματος. Εδώ βεβαίως οδηγούμαστε και στο πρώτο πρόβλημα το οποίο έχει ταυτοποιήσει η μελέτη. Ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια. Αυτό είναι μια απέτηση και ένα κεντρικό στοιχείο το οποίο ζητά η κοινωνία των ε, πολιτών. Ε, δηλαδή ε, ζητούν όλο και μεγαλύτερη λογοδοσία, όλο και, συγγνώμη, όλο και μεγαλύτερη διαφάνεια η έλλειψη διαφάνειας μπορεί να θίξει την εικόνα ε, του ε, οργάνου. Επομένως, οι δείκτες διαφάνειας δείχνουν σημαντική διασύνδεση ανάμεσα στην επίγνωση και την γνώση της εργασίας του Κοινοβουλίου αφενός και την εμπιστοσύνη που δείχνουν η κοινωνία των πολιτών, οι πολίτες προς το κοινοβουλευτικό αυτό όργανο ε, ε, σχετίζεται βεβαίως και με το περιβάλλον των εμπλεκομένων μερών. Εμείς το ε, ε, έχουμε, εκεί έχουμε βρει τρεις κατηγορίες εμπλεκομένων μερών. Το πρώτο είναι οι internal actors, οι εσωτερικοί δηλαδή ε, παίκτες, οι φορείς. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους εξωτερικούς θεσμικούς παράγοντες, δηλαδή ε, εκεί μπορούμε να αναφέρουμε τους οργανισμούς ε, λογιστικού ελέγχου, τις ιδιωτικές εταιρείες λογιστικού ελέγχου, τα Υπουργεία κτλ. Και έχουμε και την τρίτη κατηγορία που είναι οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς στην κοινωνία, οι οποίοι μπορεί να αναφέρονται ως ε, ανεξάρτητοι, μπορούν να δώσουν την εξωτερική αντικειμενική τους γνώμη προς την όλη διαδικασία και που βεβαίως μπορούν να βοηθήσουν τους ε, πολίτες ε, είτε να μελετήσουν είτε να αξιολογήσουν την κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Έχουμε λοιπόν άλλο ένα στρώμα εντός εισαγωγικών ελέγχου των δημοσίων οικονομικών. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ε, εμπλεκομένων φορέων που πραγματικά εμπλέκονται στην διαδικασία, ε, κοινοβουλευτική διαδικασία απαλλαγής εσωτερική και εξωτερική. Όσον αφορά την ίδια την διαδικασία, διαπιστώσαμε μεγάλη διαφοροποίηση των πρακτικών στα Εθνικά Κοινοβούλια. Να θα σας δώσω κάποια παραδείγματα τα οποία μπορούν ε, να ε, δείξουν τη διαφορά αυτή. Ας πούμε, να σας πω ότι η Γερμανία, στη Γερμανία το Bundestag ε, έχει μια πολύ καλή διαδικασία απαλλαγής, ε, γιατί θεωρούν ότι η καλή προετοιμασία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή περαιτέρω επιπλοκών. Σε κάποιες άλλες χώρες μέλη όμως δεν υπάρχουν έτσι, ε, τυπικές ε, διαδικασίες προετοιμασίες της απαλλαγής στην Ισπανία, ας πούμε, στην Πολωνία. Εκεί βασίζονται ε, σε εξαντλητικό εσωτερικό σύστημα monitoring που δίνει τη δυνατότητα στο θεσμικό όργανο να αξιολογήσει τους κινδύνους σε μία φάση, σε ένα στάδιο στο οποίο ακόμα μπορούν να ληφθούν διορθωτικά μέσα. Όσον αφορά την εμπλοκή των εξωτερικών θεσμικών παραγόντων, έχουμε ας πούμε την περίπτωση της Εστονίας, όπου ε, το ε, ελεγκτικό συνέδριο, το κρατικό δηλαδή όργανο, ε, προετοιμάζει την, τον προϋπολογισμό. Ε, επίσης, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούμε να αναφέρουμε, να το αναφέρουμε μάλλον σαν ε, σαφές παράδειγμα του πώς η πίεση του, των πολιτών οδήγησε σε αλλαγές. Οι δαπάνες χωρίστηκαν σε δύο αφενός λειτουργικές δαπάνες και αφετέρου δαπάνες ε, των μελών του Κοινοβουλίου. Και αυτό έγινε μετά από πίεση. Ελπίζω ότι τώρα ανέβει το μικρόφωνο του ομιλητής, ζητούμε συγγνώμη, λέει και από τώρα πήρατε μια ιδέα για το τι γίνεται όσον αφορά τις απόψεις, όσον αφορά ε, το τι κάναμε ε, όσον αφορά αυτές τις ε, περιπτώσεις, αυτές τις υποθέσεις μελέτες που αναλύσαμε και ως συμπέσμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι πιο εξαιρετικέ πρακτικέ που βρήκαμε και θα τις μπορούσαμε να συστήσουμε σαν πρακτική απαλλαγή προπολογισμών ήταν αυτές και να σταθούμε λίγο παραπάνω όσον αφορά τις συστάσεις υπαριθμών 1 και 2 και ίσως θα μπορούσα να μακρηγορήσω σε σχέση με το τι θα πρέπει να κρατήσετε από αυτή τη μελέτη. Τα εξή. Πρώτα πρώτα. Υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές. Σας τα είπε εδώ η συναδελφός μου. Και επομένω έχουμε πάρα πολλά από πλευρά αυτών των ανταλλαγών και επομένω το πιο σημαντικό είναι να ε, είμαστε εναργείς, να ε, μπορούμε να είμαστε ενημερωμένοι όσον αφορά την καθημερινή πρακτική ε, για αυτού του είδους τις ε, δαπάνες σε σχέση με τον προπολογισμό. Επίσης ε, θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτού του είδους η εξωτερική εμπλοκή δεν είναι αρκετή και η εμπλοκή των διαφορών παραγόντων. Οπότε, πρώτα πρώτα έχουμε τους θεσμικούς εμπλεκομένους που είναι κομμάτι του συστήματος σε διάφορες χώρες ας πούμε το ηλεκτρικό συνέδριο ή κάποιου ε, ανεξάρτητες ε, εξωτερικές ιδιωτικές εταιρείες ελέγχου, αλλά υπάρχει και αυτό που σας είπε η συνάδελφος, η Κάρλα, ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και όσον αφορά ε, τον, τον κόσμο, το κοινό, για να έχουν ό,τι μπορούν, για να μπορούν να αναλύσουν τα νούμερα και θα πρέπει να έτσι να κέρδισαν στην Και αυτό επίση είναι δύσκολο σαν κίνηση. Επίσης, τρίτο, θα πρέπει να έχουμε ένα στέρεο, στεγανό σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου, το οποίο να δημιουργεί εμπιστοσύνη. Και κάθε φορά που υπάρχουν επομένω κάποια ερωτηματικά σε σχέση με δαπάνε, σε σχέση με τον προπολογισμό, να μπορεί κανεί με αυτοπεποίθηση να απαντήσει και σιγουριά και αυτό διότι ε, ε, ήδη έχει κάνει τα διαβήματα τα οποία απαιτούνται. Αυτά επομένω σε τέτοιου πλαίσιο θα πρέπει να υπάρχει και πολύ, πολύ επίπεδο σύστημα. Επίση θα πρέπει όλα αυτά να τα δημιουργούμε. Με αυτά να δημιουργούμε συγγνώμη, προσβασιμότητα και διαφάνεια όσον αφορά το κοινό για τον προπολογισμό. Επίση θα πρέπει να βελτιωθεί ε, η βάση δεδομένων, η βάση το, της τεκμηρίωσης και σε πολλά κρατημέλη ανέκυψε αυτό όσον αφορά το πώς θα υπάρχει τέτοια υποχρέωση απόδοση λογαριασμών, λογοδοσία όσον αφορά τις δημοσίες δαπάνες με κάποιο ανεξάρτητο φορέα και ακριβώ όπως είπαμε έχουμε και το τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου η πίεση του κόσμου δημιουργήσε ένα τέτοιο σύστημα. Παρά το ότι βέβαια αυτό δεν άρεσε σε κάποιους κοινοβουλευτικούς αλλά εν γέννη ε, ε, ωφέλησε τα θεσμικά όργανα. Αυτό το οποίο έγινε. Επίσης, την εμπλοκή επομένω σε μια τέτοια διαδικασία απαλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, ακριβώς όπως αναφέρεται στην έκθεση, μιλήσαμε για την εμπλοκή των εξωτερικών επαγγελματιών, την συνδυασμένη ε, ε, συμβολή των θεσμικών οργάνων, την εξωτερική γνωμοδότηση. Και έτσι, ο εσωτερικό ελεγκτής θα έχει βαθμένο ρόλο και θα συνεχίσει επίσης τις συστάσεις. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ... Θα, θα δώσει μια συνέχεια τόσο πάνω στις συστάσεις που κάνει και είπαμε ότι αυτές οι συστάσεις θα πιάνουν τόπο, θα ακολουθούνται και τα επόμενα χρόνια και θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν χρήσιμο, η διαφάνεια. Σε σχέση με κάποιο είδου ετήσια έκθεση ενοποιημένη για τα σχετικά ποσά και στοιχεία, οπότε και να υπάρχει ευκαιρία και δυνατότητα να εμπλέκονται εξωτερικοί ελεγκτές και βέβαια θα πει πρέπει να παιδιά τη μετρητή αυτό το οποίο λένε. Ναι. Αλλά σίγουρα και ωφελούνται τα θεσμικά όργανα από την δημιουργία εμπιστοσύνη. Πάνω ο μιλητή, θα πρέπει να υπάρχει όμω μια βάση τεκμηρίωση και επομένω μια τυποποιημένη διαδικασία απαλλαγή ε, γνωρίζει πάρα πολλέ μορφέ και έχει μεγάλη ποικιλία από κράτο σε κράτο. Και θεωρούμε πάντως ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο το ότι μπορεί κανείς να ξέρει σε ποιο σημείο της διαδικασίας βρίσκεται όσον αφορά τον αυτοέλεγχο. Αλλού βέβαια υπάρχει διαδικασία απαλλαγή, αλλά δεν είναι τόσο τυποποιημένη, δεν προβλέπεται ρητός όπως στην Ισπανία, Τσεχία, Πολωνία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εκεί υπάρχουν παραθυράκια που μπορεί να εκμεταλλευτεί για να προβεί σε καταχρήσεις. Και τέλο πάντων θα μπορούσαμε να πούμε έτσι σαν, σαν ε, κατάληξη ότι ανοίξτε τα παράθυρα και δεν θα το μετανιώσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χάμερ, κύριε Λόπε Φερνάντε για την εισήγηση που κάνατε, για αυτή τη μελέτη που είχε συμβάσματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Βεβαίω, Φυσικά οι τον λόγο. Πρώτα πρώτα ο εισηγητή μας, ο κύριος Γκέρ Μπράντι. Σας ευχαριστώ και του δύο για αυτή την έκθεση και όντω ε, αυτό το, στο οποίο καταλήξατε στο ότι πρέπει να ανοίξουν τα παράθυρα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο συμπέρασμα κατόπιν της εκθέσεω και νομίζω ότι με αυτή τη μελέτη ε, ε, έτσι δίνεται μια όθηση ούτως ώστε και εμείς να μεταρρυθμίσουμε τη διαδικασία τη δική μας για την απαλλαγή από τον προϋπολογισμό, ε, να μπορέσουμε να, να, να, μελετήσουμε τα κοιτάπια μας και να δούμε και την ευθύνη μας όσον αφορά τις δικές μας δαπάνες. Μια ναι, που υπάρχει ολόκληρη προβληματική για το κατά πόσον το Κοινοβούλιο θα πρέπει να απαλλάσει εαυτόν. Ε, δεν υπάρχει άλλη λύση, οπότε πάρα πολύ ευχάριστο το ότι υπάρχει αυτή η μελέτη από πλευρά ε, των μελών ε, και ο Καναδά τα ίδια πράτη, αλλά έχει άλλα επίπεδα διαφάνεια. Και η σύγκριση μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν νομίζω ότι μας ε, δείχνει, δείχνει ότι έχουμε ότι υστερούμε τέλο πάντων, είμαστε κάπου στη μέση σε σχέση με το πώ έχουμε δομήσει τη διαδικασία μα απαλλαγή. Αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία σε αυτή τη μελέτη που μπορούν να μα βοηθήσουν να βελτιώσουμε την απαλλαγή. Έχω τι εξή παρατηρήσει. Πρώτα-πρώτα. Αυτό το οποίο μου άρεσε είναι σε μια τη πρώτε διαφάνεια που λέει ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία προπολογισμού. Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για μια δική μας, εσωτερική μας υπόθεση. Εδώ. Και οι ψηφοφόροι όμως βρίσκονται τελείω εκτός διαδικασίας. Τέλος πάντων, στερούνται των πληροφοριών για τη διαδικασία απαλλαγής. Το στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χάμερ είπε να ανοίξουμε τα παράθυρα, αλλά νομίζω ότι η έλλειψη διαφάνειας θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά. Έχουμε μια ματιά που στη διαδικασία, βεβαίως και έχουμε ιστορικό ελεγκτή. Όμως δεν δημοσιοποιούνται οι δικές του εκθέσεις. Απλώς ο εισηγητής συνεργάζεται στενά με τον ελεγκτή, τον οικονομικό και έχει μεγάλη σημασία αυτή η συνεργασία και πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα που εξάγονται και θα πρέπει σίγουρα και γιατί όχι να είμαστε πιο ε, καλεί στην υπόθεση τη περίπτωση διαφάνειας. Ε, πάντως παραμένει εσωτερικός έλεγχο. Επίσης υπάρχει η αιτήσια εκθέση του ελεκτικού συνεδρίου που αφορά το κοινοβούλιο και τι κάνουν. Σε λίγε γραμμές κάνουν με ένα δειγματοληπτικό έλεγχο. Ε, με τίποτα από μέσα αυτό δεν είναι έλεγχο έλεγχος των α πούμε λογιστικών μα βιβλίων. Υπάρχει όμω κάποια έλλειψη διαφάνεια στο, στο κοινοβούλιο και υπάρχουν κάποιε χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο που απεισχόλησε και την μελέτη και εκεί το ελεγκτικό συνέδριο δημοσιεύει όλο το περιεχόμενο του οικονομικού ελέγχου επί του Κοινοβουλίου. Και αυτό νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε το συζητήσουμε και Άλλο στοιχείο που το δανειζόμαστε και αυτό από τον Ηνωμένο Βασίλειο, την υπόθεση του εξωτερικού ελέγχου. Ίσως αυτό είναι κάτι που ε, δυσκολεύει πολύ κάποιους συναδελφούς αλλά, κάποιους του κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει πάντως να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί από καιρούς καιρών χρειάζεται κάποιος αμερόληπτος, ανεξάρτητος οικονομικός ελεγχτή. έχουμε. Ας πούμε να είχαμε στη, στο μέσο τη θητεία ε, ένα τέτοιο έλεγχο και έτσι να έχουμε μια βάση τέτοια εργασία και έχουμε επίση και τον ε, Καναδά που επίση και εκεί δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα. Δεν λέω όλα να δημοσιεύονται, αλλά τουλάχιστον τα μέλη της Επιτροπής μας να μπορούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα του τι γίνεται στο εσωτερικό έλεγχο. Καλύτερα από ό,τι τώρα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε. Ο ρόλος του Προέδρου είναι κάτι το οποίο δεν απασχόλησε αρκετά όσο θα έπρεπε την μελέτη. Γιατί νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα του Κοινοβουλίου να λάβει την ευθύνη του και όχι απλώς να προεδρεύει τις ολομελίες και τα σχετικά. Να αναλαμβάνει ο Πρόεδρος τις ευθύνες, να είναι υπόλογος για τις δαπάνες του Κοινοβουλίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν ρόλο, σαν αρμοδιότητα για το Κοινοβουλίο και δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν ισχύει στο δικό μας Κοινοβουλίο, γιατί προσωπικά δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της απαλλαγής. Γιατί να μην έχουμε μια δημοσία συζήτηση στην Ολομέλεια και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να συνηγορεί υπέρ των δαπανών του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πιο υπεύθυνο και δίδει και στο πρόσωπο του Πρόεδρου επίσης και στη θέση του μια υπευθυνότητα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, είναι κάτι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε μια τέτοια μελέτη Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο τη κυρία Λόπε και του κυρίου Χάμερ γιατί δεν υπάρχουν ε, πρώτερε μελέτε από αυτού. Η ερώτησή μου είναι, εσείς τι θεωρείτε, υπάρχει σοβαρή έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά την απαλλαγή. Πέραν αυτού πάντως, το να έχουμε στα κυρία μας αυτή τη μελέτη, δεν φτάνει, γιατί θα πρέπει να εξεργαστούμε τα αποτελέσματα περισσότερο. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν λόγοι βάσιμοι, ώστε να μελετήσουμε περισσότερο το θέμα. Και Πρόεδρε, εσείς θα πρέπει να το σε αυτή την ε, πρόκληση, ε, να έχουμε κάποιες ε, προτάσεις στην Επιτροπή μας. Θα μια συνέχεια σε αυτή τη σύντομη συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε με το Προεδρείο, με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Και έτσι θα να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις για το άμεσο μέλλον. Οπότε και να βελτιώσουμε σημαντικά τη διαδικασία μας χορήγησης απαλλαγής. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέρβαντη, Είμαι βέβαιος ότι πρόκειται για άλλη μια πρόταση που θα κάνει το Προεδρείο συνήθως να μας λατρέψει, να μας αγαπήσει, να μας συμπαθήσει και ξέρετε παρακολουθούν από κοντά. Άγρυπνο μάτι της ε, εργασίας μου. Τόσο αστείευαμε, έχετε δίκιο. Είναι τώρα η στιγμή να προβληματιστούμε ε, για το τι γίνεται στα κάτι μέλη, να δούμε τι κάνουν τα εθνικά κοινοβούλια. Τα εθνικά κοινοβούλια επίση να διδαχθούν από αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά πάντω να πούμε και για το τι θα κάνουμε όσον αφορά το δικό μας πρόγραμμα εργασία δική μα προσέγγιση. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας απασχολεί το θέμα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, αλλά μια που μου απευθύνατε ε, άμεσα ω πρόεδρο της Επιτροπή, θα ήθελα να σα πω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη μα για μια καλύτερη διαδικασία. Και έχω και κάποιε ερωτήσει. αλλά θέλουν να υποβάλουν πρώτα-πρώτα και άλλοι συνάδελφοι. Ερωτήσει θέλουν τον λόγο. Ο επόμενο. Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τη μελέτη. Ομολογώ ότι δεν την έχω ακόμη αναγνώσει, θα το κάνω όμως και με μεγάλη προσοχή, διότι όταν σπάνε κάποια ταμπού, τουλάχιστον πρέπει να ξέρει κανεί ποια ταμπού σπάει θα την αναγνώσω με την επιμέλεια που με διακρίνει. Να πω λίγα στον κύριο Γκερμπράντι τώρα. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν ασχολούμαστε με τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Σε σύγκριση με τον προπολογισμό δηλαδή, τη Κομισιόν, του Κοινοβουλίου τον προπολογισμό τον εξετάζουμε πολύ προσεκτικότερα. Ίσως βέβαια να μην κάνουμε πάντα τα σωστά πράγματα, διότι δεν έχουμε πάντα τι σωστέ πληροφορίε. Ίσως πρέπει να εξετάσει κανείς και τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας του κανονισμού που όπως σε κάθε κοινοβούλιο ο απλός κοινοβουλευτικός, ο απλός βουλευτής απομακρύνεται διαρκώς από, διαρκώς από τις ε, αποφάσεις. Από τότε που είμαι εγώ Ευρωβουλευτής βλέπω την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου να χάνει όλο και περισσότερο αρμοδιότητες διότι τις ανακτά το Προεδρείο. Φαίνεται λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο δεν δίνει δικαιώματα στους πολιτικούς, στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου ούτε καν. Ούτε καν οι επίτροποι δεν έχουν. Αυτό ήταν βέβαια και το θέμα της ακυρωθήσεις ακροάσεως. Να εξετάσουμε δηλαδή πόση επιρροή έχουν πραγματικά οι πολιτικοί στις αποφάσεις για τον προπολογισμό. Ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Υπάρχει η υποχρέωση υπολόγου για τους υπαλλήλους. Ο ανώτατος υπάλληλος του Κοινοβουλίου που είναι Γενικός Γραμματέας και υπογράφει τελικά τις αποφάσεις είναι υπόλογος απέναντί μας. Δεν μπορεί να υπογράφει ο πρόεδρος και να βάζει το κεφάλι του στον τορβά ο Γενικός Γραμματέας. Εμένα με απασχολεί το θέμα από τότε που έγινα εισηγήτρια του προπολογισμού το 2005, πώς θα τα καταφέρω δηλαδή, ώστε οι πολιτικοί, άντρες και γυναίκες, να έχουν περισσότερα δικαιώματα και περισσότερες υποχρώσεις επομένω για τον προπολογισμό και τις δαπάνες. Έχω μεταβεί μαζί με τον κύριο Τόιρερ και σε περιφερειακό Κοινοβούλιο και γνωρίζω το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων τι εξουσίες έχει. Για σύγκριση όμως με τα Εθνικά Κοινοβούλια βρίσκω ότι εμείς έχουμε πολύ περισσότερο ευθύνη υπολόγων εδώ. Απόδοσης λογαριασμών δηλαδή. Ούτε γνωρίζω οι Ιταλοί συνάδελφοι να έχουν προκαλέσει πρόβλημα για, την, το χτίσιμο της πισίνας στην Βουλή τους. Εμείς εδώ αεμποδίσαμε να φτιαχτεί πισίνα στην, ε, στο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, πράττουμε τα σωστά, βάζουμε τις σωστές ερωτήσεις στη διαδικασία απαλλαγή. Και οι ανεπίσημες ποιε ανεπίσημε πληροφορίε μπορείτε έστω να μα δώσετε και πού θεωρείτε ότι είμαστε καλύτεροι από τα Εθνικά Κοινοβούλια και πού είμαστε χειρότεροι σε ό,τι αφορά την διαφάνεια και σε ό,τι αφορά βέβαια την υποχρέωση απόδοση λογαριασμών. Αυτή είναι η ερώτησή μου προ του ειδικού. Υπάρχει κανεί που δεν τον πρόσεξα, λέει ο πρόεδρο. Προσθέτω και εγώ μια ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω κατά πόσον η ανάλυση των διαδικασιών ελέγχου προϋπολογισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων που κάνατε σας έχει δώσει κάποια στοιχεία κινούνται σύμφωνα με την αρχή του New Public Management. Διαπιστώνουμε εμείς ότι μέσα στα πλαίσια του ενιαυσίου του προϋπολογισμού, βράχει πρόθεσμα, δεν αλλάζει η στάση των διοικήσεων στους, ε, στις δημόσιες δαπάνες. Το μέγα μέρος ε, λοιπόν είναι δαπάνες διοικητικές οι οποίες έχουν ε, σχέση επίσης και με τις υποχρεώσεις κοινωνικών ασφαλίσεων. Είναι, είναι κόστος συντηρήσεως επενδύσεων που έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν. Έχουμε κάνει λοιπόν μεγάλες προσπάθειες ξεκινώντας στο εθνικό επίπεδο και από το επίπεδο των, των δήμων και κοινοτήτων και ανεβαίνοντα στο περιφερειακό και ούτε καθεξής, να εξετάσουμε και την προσέγγιση του κύκλου ζωής. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι στην ανάλυση, στη μελέτη που διεξαγάγατε προσέξατε να υπάρχουν κάποιες διαφορές, είδατε κάποιες best practice που δείχνουν ότι ο έλεγχος του προϋπολογισμού δεν είναι στην πραγματικότητα μόνο μια αναδρομική ανάλυση των εκθέσεων του ελεκτικού συνεδρίου, ούτε μόνο η διαπίστωση της ακριβίας των σφαλμάτων, αλλά και μια μελέτη της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, καθώς επίσης και με μια προσέγγιση προοπτικής, δηλαδή για το μέλλον. Ελπίζω ότι είναι ξεκάθαρα αυτά που ρωτώ και επίσης η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όταν πρόκειται δηλαδή για δημοσιονομικά ελλείμματα, πώς προκύπτουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και πώς μπορούν να αποφευθούν, πώς επίσης μπορούν οι χώρες να επανέλθουν στην οδό της ανάπτυξης. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις, λοιπόν αυτό ήταν το μπουκέτο των ερωτήσεων τώρα από, το, από την Επιτροπή μας. Παρακαλώ να απαντήσετε. το δεύτερο κομμάτι ήταν ε, η ίδια η μελέτη. Ναι, να μας δώσετε έτσι κάποιες ιδέες, ε, κάποια περισσότερα στοιχεία. Θα προσπαθήσω. Νομίζω ότι το ζήτημα των σωστών ερωτήσεων που πρέπει να θέσουν οι κοινοβουλευτικοί έτσι ώστε να μπορέσουν καλύτερα να ασκήσουν ε, ένα είδος πολιτικής έτσι, εποπτείας ε, επί των χρημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ε, και σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν με τον ορθότερο τρόπο σχετίζεται το ερώτημα αυτό με αυτό που είπατε δηλαδή, συνδε, δηλαδή η σύνδεση των μελλοντικών προϋπολογισμών με τον στόχο. Θέση στόχων λοιπόν ε, για το τι θέλουμε να επιτύχουμε. αλλάζει ο κόσμος και πρέπει να προσαρμοστούν και τα κοινοβούλια και πρέπει να έχουν καλύτερη στοχοθέτηση. Ένα παράδειγμα για τις δυσκολίες για τις δυσκολίες που συμβαίνουν είναι ότι ας πούμε τα μέλη της διοίκησης ε, του Κοινοβουλίου στην Γερμανία και νομίζω ότι επανερχόμενοι στο, στη διαφάνεια με το ε, διοικητικό κόστος που είναι μεγάλο στην ε, γερμανική περίπτωση εκεί λοιπόν είχαμε ένα ενδιαφέρον σχόλιο ο όγκος των χρημάτων παραμένει ίδιος, όμως υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την χρήση των χρημάτων. Ας πούμε μας είπαν ότι το θέμα της ε, ε, του μηχανισμού ας πούμε σταθερότητας απέτησε χρήση πόρων για μελέτες και για τεκμηρίωση που θα χρειάζονται οι βουλευτές. Νομίζω ότι η ο απλός οικονομικός έλεγχος, ο έλεγχος των αριθμητικών στοιχείων, έστω και αν αυτά τα στοιχεία είναι πιο σωστά, δεν δίνει την πραγματική εικόνα της σωστής κοινοβουλευτικής εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν ίσως θα πρέπει να συνδυαστούν διάφορα στοιχεία. Spending ε, ενδεχομένως δηλαδή το συνολικό ποσό να είναι ίδιο αλλά το αφήγημα που περιέχεται είναι διαφορετικό κάθε φορά. Γιατί ε, κάθε φορά υπάρχει άλλη εστίαση από πλευρά των βουλευτών. Από τις επαφές που είχα εγώ κατάλαβα ότι ε, υπάρχει μεγάλη ανάγκη πόρων για τα κοινοβούλια και στο εθνικό περιβάλλον και στα, ε, στο ευρωπαϊκό χρειάζονται χρήματα. Και ε, βεβαίως καλύτερη επεξήγηση των δραστηριοτήτων. Αλλά αυτό γίνεται καλύτερα από μέσα και όχι απ' έξω. Οι προτάσεις λοιπόν που άκουσα είναι ότι ε, πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα, πρέπει να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε καλύτερα πώς ε, ε, μπορεί να υπάρχει σταθερή κατηγορία στο εσωτερικό της οποίας όμως να λαμβάνουν χώρα πολλές τροποποιήσεις. Και κάτι άλλο το οποίο όμως δεν μελετήσαμε σε βάθος στη διάρκεια αυτής της έρευνας και εδώ μάλλον καταδεικνύεται και μία έτσι, μια έλλειψη, ένα κενό της μελέτης. Ε, ε, σχετίζεται με τη διαφάνεια. Όταν ε, εκπονείται ο προϋπολογισμός, ο οποίο δεν είναι μόνο για την επόμενη χρονιά, πρέπει να είναι λίγο πιο μακρόπνος ε, για τα επόμενα πέντε χρόνια, α πούμε, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όραμα. Εκεί, εκεί θα πρέπει ε, να έχουμε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, ένα συγκεκριμένο τρόπο διήγηση που θα έχει συνέχεια στα επόμενα πέντε χρόνια. Και σε πολλές τοπικές κυβερνήσεις βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια τέτοια τάση. Αυτά μπορώ να σας πω, τουλάχιστον σε, τούτη, σε τούτο το στάθιο. Δεν ξέρω αν η κυρία Λόπες ε, θέλει να πει κάτι σχετικά ε, με την, τα ελληπή στοιχεία όσον αφορά την απαλλαγή. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τα σχόλια που κάνατε και όσον αφορά την έλλειψη πληροφοριών για την απαλλαγή γενικά πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στο να βρούμε τις πληροφορίες αυτές. Διότι κάποια, κάποιες από τις περιπτώσεις ε, ε, μελετών των κρατών, συγκεκριμένων κρατών μιλών έχουν απαλλαγή πολύ στενή ή ε, εσωτερική, πολύ κλειστή ή εσωτερική. και είδαμε ότι η δημοσιότητα που δίνεται όχι μονάχα στους εξωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, αλλά και στις ίδιες τις διαδικασίες, δεν είναι, ε, δεν είναι πολύ εύκολη. Δηλαδή είδαμε δυσκολίες ε, συγκεκριμένες. Γι' αυτό λοιπόν χρησιμοποιήσαμε διάφορα εργαλεία και τρόπους για να βρούμε αυτά που θέλαμε. Ο καθένας έχει διαφορετική άποψη για το πώς ε, ε, εφαρμόζεται ας πούμε αυτή η διαδικασία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Θα τα σκεφτούμε όλα αυτά τα ζητήματα, να δούμε πώς ε, θα ε, εντάξουμε τα αποτελέσματα της μελέτης εργασίας μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάμερ και κύριε Λόπες Φερνάντες. Ευχαριστούμε πολύ. Τροφή για σκέψη όλα αυτά που μας είπα. Ja, ich darf dann diesen Tagesordnungspunkt abschließen und zum nächsten Ωραία λοιπόν, ολοκληρώθηκε και αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως, ήταν το σημείο 13, περνάμε λοιπόν στο επόμενο. Εκτός κι αν ο εισηγητής θέλει ξανά τον λόγο, όχι, όχι. Επομένως περνάμε στο σημείο 14 της ημερησίας διατάξεως, Στην προσωπία της Επιτροπής μας, στους λιμένες της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2012. Η Λιάννα Ιβάνοβα είναι η εισηγήτρια. Ε, θα κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, εν ώψη της ε, αποστολής αυτής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναμφισβήτητα οι λιμένες της Αμβέρσας και του Ρότερνταμ είναι πολύ σημαντικά λιμάνια. Συμμετέχουν ενεργότατα στους πόρους της ε, Ένωσης. Σκοπός της αντιπροσωπείας είναι να κάνει μια αξιολόγηση των ε, συστημάτων ε, των ε, ελέγχων στα λιμάνια αυτά. Πρώτον, δηλαδή, να κατανοήσουμε πώς στην πράξη λειτουργεί το σύστημα και επίσης πώς η φυσική επιθεώρηση καθώς επίσης και τα και πώς κρατούνται τα μητρώα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης στην και το Ρότερνταμ. Έχουμε και κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θα απευθύνομαι γιατί μας ενδιαφέρουν πολύ απαντήσεις. Ως εισηγήτρια για το θέμα του Χέρκουλ, θέλω να ακούσω από τις αρχές εάν ε, είχαν κάποια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Χέρκουλ, πώς αγόρασαν το, τον εξοπλισμό τους, τα μηχανήματά τους. Το 2010 υπήρξε, ε, έγινε η εισαγωγή του συστήματος ε, των τελωνίων χωρίς, ε, χωρίς έγγραφα, paperless customs. από ό,τι μαθαίνουμε από τις ε, εταιρείε που, χρησιμοποιούν τους λιμένες, το σύστημα δεν ε, έχει δώσει καλά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αποτελεσματικό. Ε, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί λαθρεμπόριο, παραποίηση τσιγάρων κτλ. Να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Επίσης, σύμφωνα με το υπόμνημα που έχει προετοιμάσει το τμήμα στρατηγικής δεν έχουμε ειδικέ πληροφορίες όσον αφορά ε, όσον αφορά τους εδασμούς από το Ρότερνταμ και ε, από την ε, Αμβέρσα. Ε, Ακόμα και ερχόμενοι σε άμεση επαφή με τις ε, λιμενικές αρχές και τις τελωνιακές αρχές δεν ήταν σε θέση να μας δώσουν τα στοιχεία αυτά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από τις ε, αντίστοιχες αρχές. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, σύμφωνα με τους ε, ετήσιους λογαριασμούς ε, και τις επιθεωρήσεις της Κομισιόν και τους λογιστικούς ελέγχους του 2011, υπάρχουν υπάρχουν ε, κάποιες ε, ελλείψεις στο βελγικό σύστημα διασαφήσεων ε, που σχετίζονται με τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους. Επομένως, θέλουμε αποσαφηνήσεις, διευκρινήσεις όσον αφορά τα ζητήματα αυτά. Ε, κάπως έτσι βλέπω εγώ την, τις αντιπροσωπείες στους λιμένες και του Ρότερνταμ. Ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια. ο Τίνο Έγκερμοντ της Κομισιόν και η κυρία Κλάς είναι παρόντες από τη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και από την Γενική Διεύθυνση Ταξούτ. Μπορείτε να πείτε ήδη κάτι για τις ερωτήσεις που έχει θέσει η κυρία Ιβάνοβα, πώς κρίνεται δηλαδή τα θέματα ή τι θεωρεί σημαντικό η Κομισιόν εν προκειμένου. Σε ποιον να δώσει το λόγο. Κύριε Έγκερμοντ. Να πω εγώ για το Βέλγιο που εκεί κάνω εγώ, κάνω τους ελέγχους για το όνομα της Κομισιόν. Υπάρχουν προβλήματα όντως σε ό,τι αφορά την τήρηση λογαριασμών των δασμών και αυτό διότι γίνεται κεντρικά από το 2007 σε ένα μόνο γραφείο ιτήρηση των λογαριασμών, ενώ παλαιότερα ήταν 57. Και έχουν κάνει και δηλώσεις άειλες πλέον, χωρίς χαρτιά δηλαδή, χωρίς έγγραφα. Είναι ένα νέο συνδυασμένο σύστημα, το οποίο αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, διότι δεν έγινε φάση δοκιμασιών ήταν ένα big bang δηλαδή και ξεκίνησε, κανείς δεν ήταν βέβαια έτοιμος. Εμείς κάναμε επανειλημμένα επιθεωρήσεις ήδη από το 2008. Μετά από αυτές αναθεώρησαν όλες τις πληρωμές τους μέχρι σήμερα. Ωστόσο, ακόμα αντιμετωπίζουμε δυσκολίες ό,τι αφορά την αξιοπιστία του λογιστικού του συστήματος, καθώς και για τα ποσά που μεταφέρονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γι' αυτό ζητήσαμε από τις βελικές αρχές να διεξαγάγουν εξωτερική, εξωτερικό έλεγχο για όλο το σύστημα. Πήρε χρόνο μέχρι να τους πείσουμε, εν τέλει όμως γίνεται τώρα μια πρόσκληση για υποβολή προσφορών, θα αρχίσει περίπου αρχές Οκτωβρίου, θα επιλέξουν έναν εξωτερικό σύμβουλο και θα διεξαγάγει αυτός ελέγχους σε τρεις πτυχές για τα, σύστημα, για τα συστήματα μάλλον επιστροφής. Το ποσό είναι του ύψους, του 126 εκατομμυρίων. Εμείς δεν αρνούμαστε να πληρώσουμε μέχρι να δούμε το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού. Το δεύτερο είναι για την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος και το τρίτο αναφέρεται στην έγκριση και πιστοποίηση του λογιστικού, των λογιστικών ελέγχων από εξωτερικό ελεγκτή. Ελπίζουμε η εναρκτήρια συνεδρίαση να είναι στα τέλη Οκτωβρίου και τα πρώτα αποτελέσματα να τα λάβουμε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Εδώ σας διέγραψα το πλαίσιο σε ό,τι αφορά την συλλογή και λογιστικά συστήματα. Όσον αφορά τους αποτελεσματικούς ελέγχους, εδώ πρέπει να είναι κανείς προσεκτικός με την έννοια ότι δεν είναι η περιοδικότητα και ο αριθμός των ελέγχων που έχουν σημασία. Υπάρχουν χώρες όπου έχετε μόνο 0,5% των ελέγχων. Αν όμως αυτό γίνεται σε μια καλή βάση αξιολογήσεως και με καλά προφίλ κινδύνου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτως ή άλλως αυτή είναι η γενική τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια απλοποίησης και διευκόλυνσης και ούτω καθεξής, αλλά πρέπει να είναι καλύτερη η αξιολόγηση κινδύνου. Και τονίζουμε και στις χώρες μέλη, στην χώρα μέλος, ότι η μείωση των ελέγχων στην ε, περίοδο δήλωσης των ε, εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται και στις αποθήκες των εμπόρων όταν θα έχουν δηλωθεί και περάσει τα εμπορεύματα, τα αγαθά. Ναι. Δηλαδή εννοώ στην ε, ε φάση του εκτελονισμού. Οι κάτω χώρες ήταν πρωτοπόρος ε, για να προβλέψουν την μέγιστη απλοποίηση και βέβαια το Βέλγιο αναγκάζεται να ακολουθήσει διότι αλλιώς χάνει δουλειές. Αυτές ήταν οι πρώτες μου παρατηρήσεις. Ο Πρόεδρος, κύριε Έγκερμοντ, σας ευχαριστώ. Επιθυμεί κανείς από τα μέλη να λάβει το λόγο. Ο κύριος Γκάιερ. Ίσως να μην πρόσεξα τι λέχθηκε. αλλά αυτό που ήθελα ήταν να είναι δυνατόν να εξεταστούν τα συμπεράσματα της εκθέσεως του ελεγκτικού συνεδρίου που είχαμε πέρσι στα τραπέζια μας και όπου το ελεγκτικό συνέδριο διαπιστώνει ελλείψεις και λέει ότι οι χώρες μέλη βιάζονται υπερβολικά να εφαρμόσουν τις απλοποιημένες διαδικασίες. Και αυτό προκαλεί έλλειψη ακρίβειας που αυτή με τη σειρά της βέβαια οδηγεί σε μείωση των εσόδων. Είναι σημαντικό εμείς να μην εγκύψουμε στο θέμα μόνο ως δημοσιονομικοί ελεγκτές για το πώς δαπανά δηλαδή τα χρήματά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πώς εισπράττει τα όσα της πρέπουν, τα όσα είναι δηλαδή ε, δικαιωματικά δικά της. Αν είναι δηλαδή αρκεί, επαρκής η ακρίβεια και για την διαπίστωση των εσόδων. Η ερώτηση προς την Κομισιόν έχει ως εξή. Εάν μπορεί να δηλώσει μετά από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, αν μετά από αυτό έχουν υπάρξει κάπως ξεκάθαρα αποτελέσματα. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, εάν οι απλοποιήσεις που καταρχήν μας ικανοποιούν, διότι μειώνουν τη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Εάν αυτές ωστόσο έχουν οδηγήσει σε μια έλλειψη ακρίβειας των ελέγχων. Άλλες παρατηρήσεις παρακαλώ από άλλους συναδέλφους. Όχι. Καλώς τότε η Κομισιόν παρακαλώ να απαντήσει την ερώτηση του κ. Γκάιερ. διαβάσαμε μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση όσον αφορά την απλούστευση και κατόπιν τούτου. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να προβούμε σε μια σειρά ελέγχων. Το 2009 και 2010 επισκεφθήκαμε όλα τα κράτη-μέλη και εξετάσαμε το τι στρατηγική, τι πολιτική έχουν όσον αφορά του τελωνικού ελέγχου. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση τη απλούστευση. Αυτό το οποίο κάνουν πριν ε, προβούν δηλαδή σε τέτοιου είδου ε, απλουστεύσει και είδαμε ότι ε, εν μέρει γίνεται εκ των προτέρων η μείωση. Έχουμε δηλαδή έναν προκαταρκτικό έλεγχο πριν, πριν εκχωρηθούν, πριν γίνουν οι απλουστεύσεις. Πανεπομένως, στον τόπο ελέγχου κοιτούν ποια ήταν η διαδρομή των προϊόντων, των εμπορευμάτων, αποδείξεις κλπ. Επομένως, το σύστημα μπορεί να ελεγχθεί πριν τις απλουστεύσεις. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό το οποίο ισχύει είναι και ότι εάν κανείς το παρακάνει με τις απλουστεύσεις, τότε είναι πολύ δύσκολο να επιφέρει και τελέσει τους σχετικούς ελέγχους. Και βέβαια ε, γίνονται και μετά τον εκτελονισμό έλεγχοι πρεσβεύει η Επιτροπή, ακριβώς όπως κάνουμε ε, για τους εταιρικούς φόρους. Και επομένως μπορείτε να δείτε ότι ε, μπορεί αυτό να γίνει και στα πλαίσια των ε, δασμών των ελληνικών. Οπότε έχουμε αυτούς τους ελέγχους όσον αφορά την γενική στρατηγική του ελέγχου και επίσης γίνεται απλούστευση επί τη βάση συγκεκριμένων διαδικασιών αν ε, δεν έχουμε κάποια εμπορεύματα τα οποία ε, τα εκτελονίζουν οι συναλλασσόμενοι και είπαμε ότι περισσότερη προσοχή δίνεται στους, τα, στους δασμούς anti-dumping. Πώς δηλαδή μπορούμε να αποφύγουμε το πώς θα παρακαμφθούν ε, οι έλεγχοι αυτοί. Και επομένως πώς θα δούμε τι, τι είδους κίνδυνοι ε, υπάρχουν. Και επί τέσσερα χρόνια κατά σειρά το προσοχή μας σε αυτού του είδους τους ελληνικούς ελέγχους και επί τη βάση τούτου ε, προσπαθήσαμε να προβούμε σε κάποιο είδους ε, θεματική ε, αναδόμηση στην υπηρεσία και προσπαθήσαμε επίσης να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, με 100 τόσα και πάνω από τα δύο τρίτα αυτών ε, επιλύθηκαν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τα οποία τώρα δουλεύουν σκληρά, ούτω ώστε να μπορέσει να τεθεί ένα τέρμα στην ύπαρξη αυτών των προβλημάτων. Επομένω, πολλά τα προβλήματα, αλλά πάρα πολλά από αυτά επίσης έχουν επιληθεί. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον αυτό σας καλύπτει ως απάντηση για αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, Ελιάνα Ιβάνοβη αν θέλει να κλείσει τη συζήτηση. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς ε, το να μπορέσουμε να επισκεφθούμε αυτά τα δύο λιμάνια. Οπότε και κατόπιν θα αξιολογήσουμε αυτά τα οποία είδαμε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και που τα συζητήσαμε και τώρα τελειώνει αυτή η η συζήτηση και πάμε στο επόμενο θέμα. Έχετε πεπραγμένων από την ε, αποστολή μας στην Ισπανία. Εκεί μπορέσαμε να δούμε πολύ. Δεν ήταν η πάντων η πιο εύκολη αποστολή μια που είχαμε ένα σωρό ακαθόδη να συζητήσουμε και με τις περιφέρειες και με την κεντρική κυβέρνηση. Οπότε, συνάδελφοι, Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε την έκθεση των πραγμένων. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όπως είπατε και εσείς, δεν ήταν η πιο όπως το αποστολή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Απολαυστική θα μπορούσα να πούμε, οπότε και εγώ θα ήθελα την ευκαιρία να σας πω ότι με ενδιαφέρει και η καινούργια μας αποστολή των Ιούνιο στην Ισπανία. Ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε και τους άλλους συναδέλφους και την γραμματεία που συνέβαλαν να υπάρχει κάποιο περιεχόμενο σε αυτή μας την αποστολή. Λόγω για τον βιβλίο Μεσπανία είναι ότι παίρνει ένα σωρό κονδύλια η χώρα αυτή από το 2007-2013. 35 δις ευρώ έχουν λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά για την περίοδο 2000 με 2006 η Γενική Διεύθυνση περιφερειακή πολιτική, ε, διαπίστωσε ότι υπάρχουν κάποια θέματα, κάποια προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση για το Περιφερειακό Ταμείο. Οπότε η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου αποφάσισε ότι θα αποστείλει μια διερευνητή των πραγμάτων επιτροπή στην Ισπανία φέτο. Τώρα, όσον αφορά την αποστολή, πριν φτάσουμε, ο τύπο έλεγε έρχονται αυτοί με τα σκούρα κουστούμια να μας πούν τι θα κάνουμε. Ε, καλά δεν είναι και τόσο πολλά κουστούμια, μια που πήγαν και άντρε και γυναίκε. Από κοινοβούλιο που ξεκίνησα με την Μαδρίτη, συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Πιο πολύ θύμτη μου ότι πηγή ήταν αυτή η απόφαση πάντω. Τον διαβεβαιώσαμε ότι θα ελέγξουμε. Βοήθησε όσο μπορούσε. Αυτό που θέλαμε ήταν να υπάρξουν βελτιώσει και το μέλλον. Και επίση μα διαβεβαίωσε ότι θέλει να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι όσον αφορά τη διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο. Επομένω ήταν μια ουσιαστική συνάντηση. Επίση την πρώτη μέρα συναντήσαμε τον Υπουργό των Οικονομικών και Εσωτερικών και διάφορου γενικού διευθυντέ που από τα χέρια του περνούν το κοινωτικό χρήμα. Οπότε και είπαμε ότι έχουμε τα θέματα των λεγόμενων τροποποιήσεων, ε, δηλαδή τι γίνεται, ε, πώ τροποποιούνται οι συμβάσει αφού κατακυρωθεί στο διαγωνισμό η αρχική σύμβαση. Συνεχίζεται τέλο πάντων ο διάλογο Κομισιόν και Ισπανία γι' αυτό. Επίση, η Υπουργό Μεταφορών, που επίση ε, εισπράττει πολλά την Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήσαμε τι γίνεται με κάποια άχρηστα, χρησιμοποιητά αεροδρόμια. Και έχουμε επίσης ένα σωρό ενδιάμεσους. 145 ενδιάμεση φορείς έχουν ε, επισημανθεί στην Ισπανία και αυτό βέβαια αυξάνει την πιθανότητα του λάθους. Οι Ισπανικές αρχές θεώρησαν ότι ο λόγος που υπάρχουν τόσοι πολλοί ενδιάμεσοι οργανισμοί είναι ε, λόγω της εξέλιξης της διοίκησης στην Ισπανία. Το ζήτησαμε το σε όλη την επίσκεψη. Δεύτερη μέρα. Πήγαμε στην ε, Βαλένθια με αυτό το τρένο ψηλή ταχύτητα. Ήταν από τα πιο σημαντικά σημεία τη επίσκεψη γιατί ήμασταν δίπλα στον μηχανοδηγό. Ήταν σαν, σαν να πηγαίνει κανεί στο, στο Λούνα Πάρκ. Και βέβαια η Ισπανία είναι δεύτερη στον κόσμο όσον αφορά τα τρένα ψηλής ταχύτητας. Και φυσικά πάρα πολύ κοινωτικό χρήμα έχει πέσει για αυτά τα έργα αυτών των τρένων. Εδώ με διάφορα έργα συναντήσαμε τον πρόεδρο της περιφέρειας και συζητήσαμε τα της απορρόφησης και δαπάνησης του κοινωτικού χρήματος στην περιφέρεια. Ε, Βεβαίω υπήρχε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους εκπροσώπους του τύπου, ε, οι οποίοι συνέρευσαν εκεί κατά δεκάδες και είπαμε τέλο πάντων ότι πέρα από τα λάθη προσπαθούμε να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και αυτό ήταν το μήνυμα που θέλαμε να περάσει. Μετά τη συνάντηση τύπου πήγαμε σε κάποιο πρόγραμμα για τον τουρισμό του Κοινωνικού Ταμείου Και εκεί έγινε μια αξιόλογη συζήτηση με τα μέλη της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια. Το απόγευμα επισκεφθήκαμε το Γραφείο Εμπορικών Σημάτων και την τελευταία μέρα ξαναγυρίσαμε στη Μαδρίτη. Το πρωί συναντήσαμε εκπροσώπους από Ανταλουσία και Καστήλη Λαμάντζα οι Ανδαλουσιανοί είπαν ότι τα περισσότερα λάθη πηγάζουν από ένα συγκεκριμένο ντοσιά και η Καστήλη Λαμάντζα μας είπε σε λεπτομέρειες πώς κάνουν τη διαχείριση, πώς γίνεται ο έλεγχος, ε, θεωρήθηκε ότι έχει βελτιωθεί. Επίσης, συναντήσαμε τους οικονομικούς ελεγκτές της Ισπανίας και φυσικά έγινε και άλλη μια συνέντευξη τύπου. Στις δηλώσεις μου επανέλαβα το μήνυμά μας. Και πρώτα πρώτα, πριν τη συνέντευξη που τα συζητήσαμε, θα δείτε, συνάδελφοι, την ε, ανακοίνωσή μου, τη δήλωσή μου και όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει με τους συναδέλφους και υπήρχε δηλαδή συνένεση και καλύψαμε τέλος πάντων όλα τα σημαντικά ζητήματα. Ε, η Εύα είχε κάποια θέματα, κάποια ενημέρωση έγινε όσον αφορά το, κάποια διαρθρωτικά προγράμματα, ε, διάφορες προτάσεις. Ε, πάντως, γενικά, οι συνάδελφοι συμφώνησαν ότι η έκθεσή μας αντικατοπτρίζει πιστά την επίσκεψη την αποστολή στην Ισπανία. Τους ευχαριστώ όλους που με συνόδευσαν σε αυτή την τόσο απολαυστική αποστολή στην Ισπανία. Ευχαριστώ κύριε Βόν για την έκθεση πεπραγμένων της αντιπροσωπείας. Παρόν είναι ο Γενικός Διευθυντής ή μάλλον από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής ε, δηλαδή της Κομισιόν. Έχετε το λόγο αν θέλετε για να προβείτε σε δήλωση εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Άλλος συνάδελφος πήγε στην αντιπροσωπεία αυτή, ο οποίος όμως σήμερα ασθενεί και κολλείεται. Είχαμε όμως τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα. Εμείς στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο λάβαμε και την έκθεση αντιπροσωπεία σας, γιατί η επίσκεψη αυτή ήρθε σε πολύ κατάλληλο χρόνο γιατί διαπιστώνει τις πρόοδους που έχουν γίνει μετά από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου στην Ισπανία και για τη μελλοντική περιφερειακή πολιτική. Πιστεύουμε ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην Ισπανία σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την διαχείριση των σφαλμάτων που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν. Χρειάστηκε να διακόψουμε τις πληρωμές κατ' επανάληψη διαπιστώσαμε ότι τα σφάλματα ήταν συστημικά και γενικευμένα κυρίως για τις δημόσιες προμήθειες. Τώρα όμως αναγνωρίζουμε ότι τα εναπομένα τα σφάλματα δεν είναι πλέον συστημικά. Θέσαμε το θέμα πάλι των διάμεσων, των μεσολαβούντων οργάνων, αλλά επίσης αυτό το θέμα έχει συζητηθεί. γίνεται προσπάθεια απλοποίησης του συστήματος και πιστεύουμε ότι η περίοδος 2014 έως 20 θα δώσει την ευκαιρία να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης, να μειωθούν τα μεσολαβούντα όργανα και να είναι πιο αξιόπιστες οι δραστηριότητες. Αυτά βλέπουμε από την έκθεση. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Ισπανία, μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Ε, επιθυμεί κανείς να λάβει το λόγο εκ των μελών. Η κυρία Αγιάλα. Και εγώ θα ήθελα πρώτα να μιλήσει και ο κύριος Βόνη, να δούμε τι γίνεται, ε, υπάρχουν τίποτε αλλαγές. Πρώτα-πρώτα συμφωνώ με ο κύριο Βόν υπήρχε όντως <coughs> κάποια ερωτηματικά, θα εκκρεμούσαν τα οποία έπρεπε να τα ξεδιαλύνουμε, θα έπρεπε να συζητηθεί αυτό και να διευκρινιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν έγινε αυτή η αποστολή θέλαμε να γίνει μια τέτοια έκθεση ε, κατόπιν του ε, οικονομικού ελέγχου στην Βαλένθια. Έγινε αυτή η έκθεση. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελευταία μέρα πάντως είπαμε ότι δεν προσθέσαμε όσο θέλαμε όσον αφορά τον ρόλο της, ε, του Εθνικού Ελεγκτικού Φορέα και όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δούμε πώς τα συστημικού χαρακτήρα λάθη δεν θα ξαναγίνουν. Ήταν τιτάνια προσπάθεια που καταβλήθηκε. Θα μπορούσαμε να το πούμε καλύτερα εδώ στην έκθεση, την τελευταία, στο τελευταίο, τελευταίο παράγραφο, αλλά τέλος πάντων πιέστηκαν πολύ τελευταία μέρα. Πάντως γενικά συμφωνώ. Δεν ξέρω τώρα, έχει λάβει αυτήν την ε, έκθεση οικονομικού την, την, την περιφερειακή, δεν έχει λάβει Κομισιόν. Πρέπει να μελετηθεί, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα στοιχεία που πρέπει να μελετηθούν. Έχει ζητηθεί βοήθεια λόγω οικονομικών προβλημάτων πάντως και από την περιφέρεια της ε, Βαλένθια. Επιθυμεί Άλλο μέλος, η κυρία Ορτής. Καλημέρα σας. Βεβαίως και θέλω πρώτα πρώτα να συγχαρώ την αντιπροσωπεία που πήγε στην Ισπανία. Ήταν πάρα πολύ υποδοτική αυτή η αποστολή. Εγώ νομίζω ότι θα, θα πρέπει να αλλάξουμε αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ, εκεί που αναφέρει το πρόγραμμα ε, από το Διευθυντικό Ταμείο. Αυτό δεν είναι θέμα ουσία, ήταν θέμα... Είναι, είναι θέμα διατύπωσης, γιατί συμφωνώ με το περιεχόμενο τη έκθεση. Αυτό, γι' αυτό και μόνο έχω ζητήσει αυτή την ε, αλλαγή. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο ε, έχει να κάνει το πνεύμα της έκθεσης. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Εκ των μελών, άλλος κανείς, όχι. Καλά λοιπόν, θα ρωτήσω πάλι, θα παρακαλέσω μάλλον, την ε, Κομισιόν να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Ίσως μπορεί να μιλήσει και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, λέει ο κύριος Βόν. Να απαντήσω εγώ για την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει αποκαλύψει σημαντικά, σημαντικές ελλείψεις στο παρελθόν. Φέρτε το μικρόφωνο λίγο κοντύτερα. Ωραία, ευχαριστώ. Όντως λοιπόν αποκαλύφθηκαν, όπως είπα, στην Βαλένσια το 2010 σημαντικές ελλείψεις και από την Κομισιόν και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι Ισπανικές αρχές μετά από πίεση της Κομισιόν εφήρμοσαν ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης τροποποίησης δηλαδή του συστήματος και ξανακάνοντας έλεγχο όλων των δαπανών που είχαν δηλωθεί μέχρι του σημείου που διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις. Μετά από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές λάβαμε επιβεβαιώσει ότι όλες αυτές οι ελλείψεις είχαν αντιμετωπιστεί και όλες οι διορθώσεις είχαν γίνει. Άρα επιβεβαιώνουμε τώρα ότι οι διορθώσεις αυτές ήταν ορθές. Όμως σε ό,τι αφορά δύο διαμεσολαπητικά όργανα, εξακολουθούν, οι οργανισμούς εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Ένας από τους οργανισμούς αυτός, η, ε, η, ε, η, οργανισμός της Βαλένθια για τον τουρισμό, εκεί δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα προβλήματα έχουν λυθεί. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές μας βεβαιώνουν ότι ο οργανισμός αυτός δεν, δεν θα διαχειρίζεται πλέον διαθροτικά κονδύλια. Αυτό που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εμείς λοιπόν είναι ότι δεν έχουμε λάβει ε, αξιώσεις πληρωμής από τον οργανισμό αυτό. Και σε ό,τι αφορά την ΠΙΒΑ που είναι κρατικός οργανισμός και διαχειρίζεται κρατικές ενισχύσεις, εξακολουθούν τα προβλήματα. Επομένως η ελεγκτική αρχή δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι όλα έχουν αντιμετωπιστεί, όλες οι ελλείψεις έχουν αντιμετωπιστεί, αλλά και αυτοί μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχουν δηλώσει καμία δαπάνη στην Κομισιόν μετά από την αποκάλυψη των σφαλμάτων. Έτσι η Κομισιόν δεν θα πληρώσει μέχρι σότου η ελεγκτική αρχή να δηλώσει και να βεβαιώσει ότι έχουν εφαρμοστεί όλες οι διορθώσεις. Επειδή η AVT δεν πρόκειται Εμεί παρακολουθούμε, μάλλον, ε, παρακολουθούμε την εξέλιξη με τον οργανισμό αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βον ζήτησε να γίνει και μια δήλωση από την Γενική Διεύθυνση ε, Απασχόλησης. Μπορούμε να έχουμε μια τέτοια δήλωση. Όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης το 2010, είχαμε 13 επιχειρησιακά προγράμματα στο αποθηματικό. Το 2011 από τα, ε, είχαμε 22 επιχειρησιακά προγράμματα. Εν τω μεταξύ έχει εκπονηθεί σχέδιο δράσης ε, που όμως δεν βελτίωσε πολύ το σύστημα στην Ισπανία εμείς είχαμε πει στην αντιπροσωπεία πως ε, είχε η κατάσταση όσον αφορά τις ε, διακοπές και τις ανακλήσεις ε, και να πούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα με, με κάποιες διακοπές όσον αφορά ενδιάμεσα όργανα ενώ όσον αφορά το άλλο κύριο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Λούτσα, έχουμε μερική διακοπή σε ένα ενδιάμεσο οργανισμό. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι εν συγκρίση με άλλα προηγούμενα χρόνια έχουμε σαφή βελτίωση, διαπιστώνουμε σαφή βελτίωση. the state of play at the moment. Έτσι έχουν τα πράγματα για την ώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. θα ήθελα να δώσω πάλι τον λόγο στον Ντέρεκ Βόν για να συνοψίσει. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ την Εύα πρώτα για την διευκρίνηση της σύστασης που κάναμε. Θα δω αν μπορώ να την περιλάβω στην έκθεση. Ευχαριστώ και τους άλλους συναδέλφους για τις ερωτήσεις και την Κομισιόν για τις απαντήσεις. Σημαντικό είναι η Κομισιόν να επιβεβαιώσει τα όσα βρήκαμε στην αντιπροσωπεία την ίδια τον Ιούνιο, δηλαδή ορισμένες ελλείψεις, ορισμένα προβλήματα με τα διαχειριστικά συστήματα, ωστόσο έχουν γίνει βελτιώσεις, τα πράγματα ασφαλώς είναι καλύτερα, βέβαια από την άλλη μεριά πάντα υπάρχει χώρος και για περαιτέρω βελτιώσεις. Αυτά διαπιστώσαμε την αντιπροσωπεία όταν μεταβήκαμε στην Ισπανία τον Ιούνιο. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ όλες και όλους που συμμετέσχουν στην αντιπροσωπεία. Ήταν σημαντικό που ακούσαμε αυτό το follow-up και μπορούμε να συζητήσουμε στην Επιτροπή μας γενικότερα κάπως τι θα κάνουμε για την κοινή διαχείριση διαρθωτικών και άλλων ταμείων και κάτι που πετύχαμε στο δημοσιονομικό κανονισμό αυτά που πετύχαμε μάλλον με το δημοσιονομικό κανονισμό θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει καλύτερα την διαχείριση στις χώρες μέλη. Βέβαια, την κύρια ευθύνη εξακολουθούν να φέρουν οι χώρες μέλη και οι περιφέρειές των. Ευχαριστώ και εδώ λίγη συζήτηση του θέματος αυτού. Έτσι φτάσαμε στο τέλος του, της συνεδριάσεως μας. Ευχαριστώ όλες και όλους. Ε, ήταν ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση. Ευχαριστώ και τους μεταφραστάς, καθώς και την γραμματεία της δημόσιας συνεδρίασης. Κλείνει η συνεδρίαση εδώ και παρακαλώ τους συντονιστές να μείνουν εδώ. Ευχαριστώ. Σεφ, Okay, um, dear colleagues, uh, dear co αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συντονιστές. Να δούμε αν μπορούν, μπορούν να έρθουν όλοι. Ε,